Colleagues, my apologies for falling into Paulo Costa's habits of turning up late. Μέχρι να βλέπετε ότι τηρούνται οι παλιέ ε, κοινοβουλευτικέ παραδόσει, να ερχόμαστε αργά και με την άδειά σα τώρα θα πρέπει τώρα να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει πρώτο-πρώτο, δηλαδή να κάνουμε τι ψηφοφορίε, την ψηφοφορία που γίνεται από κοινού με την ΙΜΚΟ. ΙΜΚΟ, ΙΜΚΟ. Ναι, ναι, Μάρκο, έτσι είναι το σωστό. Θέλουν όμως οι τεχνικοί μας πέντε λεπτά, ούτω ώστε να ρυθμίσουν τα μηχανήματα. Οπότε στο μεταξύ να σας πω τις ανακοινώσεις του Προέδρου. Και την ψηφοφορία λοιπόν για την ηλεκτρονική κλίση. Έχουμε την... τον κατάλογο. Οι άλλοι την έχουν, εγώ δεν την έχω, βλέπω. Ευχαριστώ το ΕΛΚ. I'll do a check anyway. Um, okay. Can we first of all do a, a check on the, on the vote? πρώτα, να κάνουμε μια δοκιμή. Τώρα ψηφίζουμε, ψηφίστε. God knows. No, it's the other way, I think. The system works. We could stop it. Okay. We haven't got anybody overvoting or whatever. Now, who... Όλα καλά. Ποιο δεν τα κατάφερε να ψηφίσει. Ποιο δεν έχει την κάρτα ψηφορίας. Μόνο ένας. Μην κάνετε πότε θα μα το λέτε. Κάθε φορά. Εκθεσιδίας πρωτοβουλίας, ηλεκτρονική ψηφοφορία, πρώτη παράγραφος, συμβαστική υπαριθμόν 1. Υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 37, υπέρ, κατά, αποχέ, απορρίπτεται, 35, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική υπαριθμών 2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για τη δεύτερη συμβαστική ψηφίζουμε Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 34-26 εγκρίνεται. Επόμενη. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 42. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική υπερθμόν 3. Υπέρ. Κατά. Απογές. Εγκρίνεται. επόμενη έχουμε μια πρόταση για προφορική τροπολογία. <coughs> Με την προφορική τροπολογία, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Αυτό είναι το 50. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτονται. 52 υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53. Υπάρχει προφορική τροπολογία. Αντιρρήσει όχι, Μας με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 4. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. 58. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 67. Υπέρ κατά αποχές Σε 69 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές ξανά υπέρ κατά αποχές Το τώρα το βλέπω ήδη έχει κουράσει 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 Περ, κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 81. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ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 κατά αποχές εγκρίνεται 102 περ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 έχει αποσυρθεί 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 όχι, 113 κάνω. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113, υπέρ, κατά, αποχές. 114, 115, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική, 14. Υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 120. Όχι. Έχει καταπέσει λόγω της συμβαστικής 3. 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές έλεγχος και το 127 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 28, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε στη συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά συγγνώμη το 7 ήταν έκανα λάθος λέει ο πρόεδρος ένα λόγο, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε για το 8 ψήφισαν όλοι Πέρας. Και εγκρίνεται 9. Πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10. πρώτη ψηφορία, πρώτα πρώτα χωρίς τη λέξη ευρύς και το δεύτερο έχει τη λέξη ε, broad, ευρύς. Στο 10 λοιπόν, χωρί τη λέξη abroad, abroad στο εξωτερικό. Abroad στο εξωτερικό. Abroad στο εξωτερικό. Και τώρα έχουμε τη λέξη abroad στο εξωτερικό. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Έντεκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 17 18 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 είναι γλωσσικό το θέμα που και έχουμε τώρα τη συμβαστική 19 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 26 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρα ψηφοφορίας 58 4 με 8 αποχές εγκρίνεται Συγχαρητήρια κυρία Συναλόβα. Και κύριε Κο, κύριε Χάρμπορ. Κύριε Χάρμπορ, πρόεδρε και θέση. Εκ μέρους της Επιτροπής Ιστορικής Αγοράς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μπράιν Σίμψον και τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών και Καφές. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ επιτυχή η συνεργασία μας και νομίζω ότι πάρα πολύ επικοδομητικά μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και είναι πάρα πολύ ωραίο θέαμα να είναι τόσοι πολλοί συνάδελφοι και να ψηφίζουν. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ελπίζω ότι στο μέλλον επίση θα επανελθεί η συνεργασία μα. Ευχαριστούμε. Και περιμένω πω και πώ να δω του συναδέλφου τη Δική μου επιτροπή ε, αύριο και την Πέμπτη. Βλέπω πολλοί φεύγουν, όχι επειδή δεν ενδιαφέρονται, αλλά διότι θα πρέπει να ετοιμαστούμε για την αυριανή συνάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Μάλκον και επίσης πρέπει να αποδίδουμε και καλή τύχη με όσον αφορά τη δουλειά σας αύριο. Ευχαριστούμε και πάλι. Okay, Tran team, don't go away. Tran team. Ωραία. Παρακαλώ την ε, Επιτροπή Τραν ε, να μην ε, αποχωρήσει, να αναφερθώ στην ε, συνάντηση των συντονιστών και τις αποφάσεις που ελήφθησαν. Σας παρακαλώ οποιαδήποτε άλλη συζήτηση να γίνει εκτός της αιθούσης.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 Thank Ανακοινώσεις του Προέδρου από τη συνάντηση των συντονιστών. Καταρχήν όσον αφορά τον ορισμό των εισηγητών. Έχουμε ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα τέλη υποδομών. Η σύσταση των συντονιστών είναι να ζητήσουμε την άδεια να ετοιμάσουμε έκθεση πρωτοβουλίας πάνω στην ανακοίνωση αυτή και να το συνδέσουμε αυτό με την πρόταση για τα ηλεκτρονικά διόδια. Θα εκπονήσουμε λοιπόν έκθεση πρωτοβουλίας που θα συνδέει το θέμα αυτό με την άλλη πρόταση της Επιτροπής. όσον αφορά τον ε, εξοπλισμό οχημάτων και τις ε, πρωτοβουλίες ε, τις, τις πρωτοβουλίες κοινών τεχνολογιών, την Τράπεζα Ανάπτυξης, 5 τα προγράμματα ανάπτυξης, 6 την απόφαση του Συμβουλίου που τροποποιεί την παράλληλη συμφωνία για ε, οχήματα, 7 όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ, 8 το πρωτόκολλο για τη Συμφωνία Ευρώπης Μεσογείου. Ε, εδώ έχουμε αποφασίσει να μην αναλάβουμε καμία δράση. Εννέα, έχουμε ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την έκθεση της πολιτικής ανταγωνισμού 2011. Ε, η απόφαση είναι να εκπονήσουμε γνωμοδότηση, ε, την οποία θα αναλάβει η ομάδα ECR. Για τα 10, 11 και 12... Ε, του βουλευτή Σέζιο Σιλβέστρης. Η απόφαση ήταν να μην αναλάβουμε καμία άμεση δράση, αλλά να φροντίσουμε το ψήφισμα να ληφθεί υπόψη στις επόμενες εκθέσεις μας για τα θέματα αυτά. Όσον αφορά το 13, τη συμφωνία με τη Μολδαβία, καμία δράση. 14, ε, κείμενο της ε, Επιτροπής ε, Κατευθυντήρες Γραμμές, πάλι καμία δράση. 15, Ανατολική Εταιρική Σχέση, καμία δράση. Το 16 επίσης. 17, αύξηση της εμπιστοσύνη ε, των καταναλωτών καμία δράση και 18 γνωμοδότηση για το πρόγραμμα σύγκλησης της Βουλγαρίας πάλι καμία δράση. Δεν θα αναλάβουμε. Έχει κανείς παρατηρήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά. Τρεις μήνες με μόνο δύο θέματα προς ενημέρωση και τον επόμενο μήνα έχουμε 19 θέματα. Ομάδα κρούσης για τον τουρισμό. Η απόφαση είναι η ομάδα να συγκροτείται από πέντε άτομα από, ε, τους, ε, από το ΕΛΚ, τρεις από τους ε, και δημοκράτες ε, και έναν από το, της από τις άλλες ομάδες. Αυτό δεν εμποδίζει κανένα άλλο μέλος του Κοινοβουλίου να συμμετάσχει στις συναντήσεις αυτές. Αλλά επειδή μας ε, ανέθεσε η Ολομέλεια να δημιουργήσουμε μια τέτοια ομάδα, ε, γι' αυτό αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη σύνθεσή της. Θα προεδρεύσει ο Πρόεδρος και ο μόνιμος εισηγητής, ο κύριος Φιντάνσα, θα είναι αντιπρόεδρος, έτσι το ΕΛΚ θα έχει ακόμα τέσσερις θέσεις. Οι συναντήσεις θα αποτελούν επίσημα μέρος ε, των ε, συνεδριάσεων της ε, ΤΡΑΝ και αν είναι απαραίτητο θα υπάρχουν περαιτέρω συνεδριάσεις χρησιμοποιώντας τις γλώσσες που έχουμε στη διάθεσή μας. Εάν δεν γίνονται στα πλαίσια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Μεταφορών οι συναντήσεις αυτές, το πρόβλημά μας είναι η διαρμηνία. Σας παρακαλώ λοιπόν ε, να το γνωρίζετε αυτό ότι θα είναι περιορισμένε δυνατότητε για τη ερμηνεία σε περίπτωση που δεν γίνονται στο πλαίσιο των συνεδριάσεων ε, της ε, ΤΡΑΝ οι συνεδριάσεις αυτές. Μετά τις 28 Ιουνίου θα γίνει η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας αυτής και θα εξετάσουμε ο κύριος Φιντάνσα και εγώ θα εξετάσουμε το πρόγραμμα εργασιών ε, μαζί με τους επίσημους βουλευτές. Αυτή λοιπόν είναι η ομάδα κρούσης για τον τουρισμό. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Οι συντονιστές ε, συζήτησαν ε, τα Τέντη και συμφώνησαν πάνω σε ένα χρονοδιάγραμμα ως εξής. δεν ε, θα γίνουν ε, δεκτές άλλες ε, τροποποιήσεις. Προθεσμία για μετάφραση της έκθεσης είναι 5 Ιουλίου του 2012. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης 6 Σεπτεμβρίου. Προθεσμία για τροπολογίες 28 Σεπτεμβρίου. Εξέταση των τροπολογιών 5 Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Τράνη 27 Νοεμβρίου και ολομέλεια τον Ιανουάριο του 2013 για τα ΣΕΦ, διότι θα πρέπει να το κάνουμε αυτό μαζί με την Επιτροπή Ίντρα. Ε, προθεσμία για μετάφραση είναι 5 Ιουλίου, εξέταση της, ε, του σχεδίου έκθεσης 18 Σεπτεμβρίου, προθεσμία για τις τροπολογίες 4 Οκτωβρίου, εξέταση των τροπολογιών 5 Νοεμβρίου, ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν 27 Νοεμβρίου και πάλι ολομέλεια ε, τον Ιανουάριο του 2013. Είστε όλοι ικανοποιημένοι με το χρονοδιάγραμμα αυτό. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πέντε, τα μεγάλα φορτηγά. Έγινε συζήτηση με τους συντονιστές ε, όσον αφορά την απόφαση του Αντιπροέδρου Κάλλας να εμείνει στην αρχική του θέση όσον αφορά το θέμα των μεγάλων φορτηγών. Ομόφωνη απόφαση των συντονιστών ήταν ο Πρόεδρος ε, να στείλει επιστολή στον Πρόεδρο Σούλς ε, εκφράζοντα την ανησυχία του σχετικά με τη διαδικασία που υιοθετεί η Επιτροπή η οποία στερεί από το Κοινοβούλιο τα ε, δικαιώματά του και δημιουργεί νομική αβεβαιότητα. Η επιστολή θα προτείνει επίσης να παραπευθεί το θέμα στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων για να ξεκαθαριστεί το θέμα και να δει τι δράση μπορεί να αναλάβει το Κοινοβούλιο στο θέμα των μεγάλων φορτηγών όλα αυτά. Ε, το φυλάδιο για την επιτροπολογία διανεμήθηκε και στα διάφορα η κυρία Λίχτενπεργκερ αναφέρθηκε και στην συνάντηση 9ης, 10ης και 11ης Ιουνίου για τον διατλαντικό διάλογο που πραγματοποιήθηκε στην Κοπενχάγη. Ευχαριστώ την κυρία Λίχτεμπεργκερ ε, που ε, συμμετείχε κατά την απουσία μου. Ευχαριστώ Εύα. Και τέθηκε το θέμα πάλι των, ε, των ε, ταχύμετρων. Θα, θα εξετάσουμε και την Ολομέλεια του Ιουλίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις σχετικά με ε, την συνεδρία των συντονιστών. Εάν όχι, μπορούμε να εγκρίνουμε τις αποφάσεις αυτές. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα στις ψηφοφορίες μας. Θα πρέπει, έχουμε την αναδιατύπωση για τους σιδηροδρόμους τώρα. The uh, single European railway area, Mrs. Serikiani's έκθεση της κυρίας Σαρικιάνη για τον ενιαίο χώρο σιδηροδρόμων. Ε, να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις στις 13 Ιουνίου, στον τελευταίο τριμερή διάλογο ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή, η τελική συμφωνία σχετικά με την αναδιατύπωση του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων. Αυτό ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο. και να πω ότι πολύ σκληρή δουλειά έκαναν και οι σκιώδεις εισηγητές ε, μαζί με τον εισηγητή. Ε, τους ευχαριστώ λοιπόν όλους. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό από, από, ε, για το Κοινοβούλιο. Ε, βλέπουμε τη δημιουργία δικτύου ρυθμιστικών οργάνων σε όλη την Ευρώπη οι υπηρεσίε που συνδέονται με του σιδηροδρόμου θα είναι πιο ανοιχτές σε όλους τους οικονομικούς φορείς και η χρηματοδότηση των υποδομών έχει διασαφινιστεί. Υπάρχει μία ρήτρα που ζητάει από την Κομισιόν να υποβάλει νομοθετικέ προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση υποδομών στις μεταφορές και σχετικά με το άνοιγμα των εθνικών αγορών επιβατικών μεταφορών και επίσης θα πρέπει να γίνουν ε, όλες οι διαδικασίες πιο διαφανείς. Πρόκειται για κάτι παραπάνω από μια κλασική διαδικασία αναδιατύπωση. Ε, βλέπουμε ουσιαστική βελτίωση του κειμένου και διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων. Η ε, ΚΟΡΠΕΡ 2 θα συναντηθεί στις 15 Ιουνίου. Περιμένουμε επιστολή που να ε, μας διαβεβαιώνει σχετικά με την βούληση της, του Συμβουλίου να υιοθετήσει το ε, πακέτο αυτό και ε, το κείμενο όπως θα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο θα ψηφιστεί στις 15 Ιουλίου. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τους σιδηροδρόμους. Ο κύριος Ρώση, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, το ΕΛΚΕ έχει θυμίσει στο Συμβούλιο την πολωνική εξαίρεση. Θα θέλαμε επίλυση του προβλήματος αυτού σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Ε, λύθηκε το θέμα, ήταν μέρος των διαπραγματεύσεων. Ο Μάικλ. Ε, αν μετακινηθεί το Συμβούλιο, τότε μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αυτή ήταν η θέση του Κοινοβουλίου. Ωραία. Ο Ρόπερτ. Ε, αν μετακινείται το Συμβούλιο, νομίζω ότι θα είναι σοφό να ακολουθήσουμε την παρέκκληση του άρθρου 17. Είναι το ίδιο πρόβλημα λίγο πολύ ή είναι διαφορετική νομική θέση. Στο σημείο 10 που είχατε συμπεριλάβει κύριε Πρόεδρε στην ε, επιστολή σας ε, θα ήθελα να επανέλθουμε. Ε, μη βιαζόμαστε, ας περιμένουμε να δούμε τι θα μας πει το Συμβούλιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι το Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο με το, τη συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας ε, στο Στρασβούργο. Όταν επανέλθει το Συμβούλιο θα πρέπει να αντιδράσουμε ανάλογα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να επανέλθω σε αυτή την επιλογή της Πολωνίας να μην συμμετέχει, θα ήθελα να αποσαφώσω ότι ότι πρόκειται για απολύτη ε, αδιαφορία για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχει διαγραφεί από την αρχή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει παραβλεφθεί και θεωρώ, και θεωρώ τη θέση μας, ε, τα δικά μας συμπεράσματα, δικές μας συζητήσεις και δικές μας αποφάσεις απλά δεν ελήφθηκαν σαν υπόψη. Έχω την εντύπωση μάλιστα ώστε στο πλαίσιο αυτού του δίθεν συμβιβασμού. Μας έχουν πει να ε, ακολουθήσουμε τη γραμμή του στο κοινοβούλιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται έτσι είναι θέμα αρχής και πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά από ότι πριν από 20 χρόνια τέτοιου είδους συμβιβασμού. όταν πριν από 20 χρόνια όλα επεβάλλονταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα όσον αφορά αυτό το ζήτημα Ξέρω ότι είναι και θέμα πολιτικής από πλευρά του Συμβουλίου, αλλά θα πρέπει να μην το επιτρέψουμε αυτό. Ε, είχαμε την πολυνική, λοιπόν, έχουμε τις πολιτικές παρεμβάσεις, κύριο Σασάντε. Να ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια αυτή η τροπολογία είχε 432 ψήφους υπέρ και στην τελευταία ψηφοφορία στην Επιτροπή Τραν αυτή η τροποπολογία είχε μόνο 13 ψήφους κατά. Η μεγάλη πλειοψηφία δηλαδή των ε, βουλευτών πλήρως, ε, ψήφισαν υπέρ αυτής της τροπολογίας. Ελάχιστη ήταν κατά και θα σας ενημερώσω ότι εμείς δεν πρόκειται να καθίσουμε να περιμένουμε να μας πει το Συμβούλιο τι έχει να πει θα έχουμε τη δική μας τροπολογία για τη δεύτερη ανάγνωση και τη δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Τράσβουργο Ευχαριστώ. Κύριε Ζάνκε. Όπως και οι συναδελφοί μου, θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προηγούμενους ομιλητές. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση. Τι νόημα έχει να ψηφίζουμε εδώ πέρα εάν το αποτέλεσμα πρόκειται να είναι διαφορετικό στην ψηφοφορία από ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Μεγάλη πλειοψηφία ήταν υπέρ αυτή τη τροπολογία. Θεωρώ λοιπόν ότι οι αποφάσει και τα συμπεράσματά μα θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά. Θέλω να συμφωνήσω με του συναδέλφου, του προηγούμενου ομιλητέ. Ευχαριστώ μάλιστα. Όπω φαίνεται, θα χρειαστεί εγώ να υπερασπιστώ την ομάδα που διεξήγαγε όλε τι διαπραγματεύσει και ούτω θα πράξω. Όταν περάσετε σε τριμερή διάλογο και σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο χρησιμοποιούμε τη δεύτερη ανάγνωση ως βάση. Έτσι κάναμε εμείς και ως Κοινοβούλιο πρόβαλαμε τις ε, εξαιρέσεις, ε, όχι απλά τις πολωνικές, αλλά και υπήρχαν και τομείς ε, που σχετίζονται με τις χώρες της Βαλτικής και την Ουγγαρία. Εν τέλει, όταν μας ρώτησαν, όταν ρωτήσαμε κατά πόσο το Συμβούλιο υποστηρίζει την επιλογή μη συμμετοχή τη Πολωνία, το Συμβούλιο απάντησε ότι κανεί άλλο δεν το υποστηρίζει εκτό από του Πολωνού. και το Συμβούλιο ε, ήταν ε, δεν το συζήτησε στο πλαίσιο αυτό της συζήτησης της όλης της αναδιατύπωσης η Κομισιόν υπέβαλε μια, ένα συμβιβασμό. Ο συμβιβασμό ήταν ότι η εξαίρεση θα μπορούσε να παραμείνει έως ότου κάποιος θελήσει να ανταγωνιστεί σε αυτό ε, το δρομολόγιο. Συνεπώς η εξαίρεση μπορεί να παραμείνει εκτός αν κάποιος δηλώσει ότι θέλει να ανταγωνιστεί σε αυτό το δρομολόγιο. Η πολωνική αντιπροσωπεία, η μόνιμη αντιπροσωπεία της Πολωνίας απέρριψε αυτό το συμβιβασμό. Εγώ θεωρώ ότι ήταν λάθος τους, αλλά αυτή ήταν η απόφασή τους. Προσπαθούμε τώρα δηλαδή να έχουμε μια δέσμη μέτρων με μια συμφωνία και ένα από τα εμπόδια θα είναι αυτές οι εξαιρέσεις. Η διαπραγματευτική ομάδα ε, δαπάνησε πέντε ώρες αποφασίζοντας ότι στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων θα απέριπτε την εξαίρεση για την Πολωνία. Οι χώρες της Βαλτικής συμφώνησαν να περάσει από άρθρο σε εκτιμώντας τροπολογίες του κ. Ζήλερ και χρειάστηκε λοιπόν να μετακινηθούμε σε διάφορα πράγματα και διάφορες επιλογές. Γνωρίζαμε τη θέση του Κοινοβουλίου για αυτό, αλλά αποφασίσαμε, όλη η ομάδα, όλοι οι σκιώδεις, αποφάσισαμε μαζί ότι θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να ψηφίσει για αυτό τον Ιούλιο. Αν λοιπόν τα μέλη από την Πολωνία δεν είναι ικανοποιημένα, τι να κάνουμε. Το ΕΛΚ ε, υπεράσπισε πολύ ισχυρά τη θέση σε εκείνη τη συνεδρίαση, αλλά μια πλειοψηφία είπε ότι πρέπει να το αφήσουμε. Φυσικά κύριε Σασάντα, έχετε όλα τα μέλη από την Πολωνία, έχετε απολύτως το δικαίωμα να ψηφίσετε κατά στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Θα δούμε τι θα συμβεί τότε. Αλλά από μέρος μου εγώ πρέπει να σας αναφέρω τι, ποια ήταν η συμφωνία τελικά με το Συμβούλιο, τι θα δεχθεί το Συμβούλιο. Και έτσι θα πράξω, έτσι έπραξα και έτσι και θα πράξω και προσπάθησα να είμαι όσο πιο δίκαιος ήταν δυνατό. Συζήτησα με τους κοιόδης συζητητές ε, και η συμφωνία είναι ικανοποιητική. Το μόνο που πρέπει να σας πω είναι ότι κάποιες στιγμές δεν μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Και σίγουρα δεν έχουμε τα πάντα στην προκειμένη περίπτωση από την άψη του Κοινοβουλίου. Αλλά κάποιε φορέ χρειάζεται να κάνει κανεί διαπραγμάτευση και άλλε φορέ χρειάζεται να υποχωρήσει. Κατά την άποψή μου, για να επιτύχουμε τη συμφωνία και με αυτό συμφωνούσαν και οι υπόλοιποι. Μια πλήρη συμφωνία για όλα τα υπόλοιπα που θέλαμε, τη διαφάνεια και όλα αυτά. Χρειάστηκε να θυσιάσουμε αυτό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν θέλω να μπούμε σε εκτενείς συζητήσει, διότι μπορούμε να το κάνουμε και στην Ολομέλεια. Ακούστηκε ότι στο Συμβούλιο η Πολωνία είπε ότι άσχετα από το, το αν υπάρχει αυτή η ρήτρα παρέκκληση ε, θα καταψηφίσουν την αναδιατύπωση. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν αυτογκόλ. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να στηρίξουμε μια τέτοια θέση. Σωστή η παρατηρήση σου, Μάικλ. Δεν ξέραμε ότι οι Πολωνίοι πρόκειται να ψηφίσουν υπέρ. Ο κύριος ε, Ich glaube, das ist unser Problem, dass wir... Νομίζω ότι το πρόβλημα μας είναι ότι δεν λαμβάνουμε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται μέσα στο Συμβούλιο ώστε να έχουμε σαφές μήνυμα. Δεν νομίζω ότι η πολωνική αντιπροσωπεία θα καταψηφίσει την αναδιατύπωση. Όσον αφορά αυτήν την παρέκκληση, που έχει να κάνει με αυτήν την ε, μία γραμμή μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμβασμού ενδεχομένως, ε, μπορεί να μην είναι ε, να μην ισχύει επάπειρο, να βάλουμε χρονικό περιορισμό για την παρεκκλησία αυτή. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση, αλλά η Κομισιόν ήταν κατά αυτού. Ε, είπαν ότι η πολωνική αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο δεν έχει μετακινηθεί καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε ε, έναν συμβιβασμό. Και σε αυτή τη θέση εμένω. Ωραία λοιπόν, επιβεβαιώνω ο κ. Κουντέκ το υπερασπίζεται μέχρι τέλους, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Οι κανόνες επιτρέπουν στους πολλούς συναδέλφους να το συζητήσουν αυτό ξανά στην Ολομέλεια εφόσον το επιθυμούν. Εγώ ως Πρόεδρος Επιτροπής ε, θα πρέπει να σεβαστώ τις διαπραγματεύσεις και την αποφάση πλειοψηφία των σκιωδών με την παρουσία μου. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφουμε στις ψηφοφορίες τώρα we have the minister coming as well, don't forget. Ε, μην ξεχνάτε ότι κάποιοι από εμά πρέπει να πάμε στη συνεδρίαση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μπορούμε να ξαναελέγξουμε για τις ψηφοφορίες, διότι έγινε επανεκκίνηση του συστήματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Everybody voted. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν άπαντες. Κλείνει η ψηφοφορία. Έχουμε έναν παραπάνω. Μάλιστα. Ε, απλά σας ενημέρωσα ότι είχαμε έναν παραπάνω. Ας περάσουμε στην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 αποχές εγκρίνεται 45 με την προφορική τροπολογία του κ. υπάρχει αντίρρηση για την προφορική τροπολογία αν όχι υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε ηλεκτρονικά τροπολογία 45 με την προφορική τροπολογία άρχεται ψηφοφορία ο ψήφισαν άπαντες κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται 51 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 5 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται 52 με προφορική τροπολογία. Αντιρρήσεις για την ε, προφορική τροπολογία. Α, καταπίπτει λόγω της τροπολογίας 6, συγγνώμη. 7 λοιπόν τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 τροπολογία 9 και 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 54 του κυρίου Τέιλερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 56 παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται 57 και 58 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκριν, απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όλες οι υπόλοιπες 24, 10, 11, 12, 13 έχουν αποσυρθεί. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της λίστας ψηφοφορίας. Συμβιβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο μέρος 3. Μου λέει ο Πίτερ, αυτό απαντάει και την ερώτησή σας. Είναι βήμα 3 ή μέρος 3. Ωραία λοιπόν. Τμήμα 3 της λίστας ψηφοφορίας, στη σελίδα 14 στο δικό μου έγγραφο, δεν είμαι... Δεν είναι η ίδια σελίδα στο ΕΛΚ. Θα είναι κάπου στο 13, 14, 15 σελίδα μάλλον. Τροπολογία 72 ουσιαστικά της κυρίας Αβισάρ. Σελίδα 13 στο ΕΛΚ, 14 στους σοσιαλιστές, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες ομάδες. Το έχουμε μπροστά μας όλοι. Παράρτημα 6, σημείο 3, παραγραφός 2, κυρία Σαββισάρ, τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, απορρίπτεται. 14 τροπολογία, διπλή ψηφοφορία σε δύο μέρη, πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, δεύτερο μέρος το υπόλοιπο της τροπολογίας υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. apparently... Όπω φαίνεται να τώρα στη συμβιβαστική 2. Είναι κατάμαυρο το κελί του πίνακα στη σελίδα μου. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 22 στη συνέχεια υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 τροπολογία υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες κλείνει η ψηφοφορία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 κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ξεκινάει η ψηφοφορία Σαν everybody voted, πέρας ψηφοφορίας, 42 υπέρ, 30 κατά, εγκρίνεται συγχαρητήρια στον κύριο Παρνιού τον εισηγητή. Now we come to Michael's three opinions. Περνάμε στις τρεις νομοδοτήσεις του Μάικλ. Πρέπει να αλλάξουμε βάρδια εδώ πάνω. Α, νάτος. Ωραία. Πρώτη είναι η γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερικής Ανάπτυξης, ε, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής που ανακαλούν ε, τον κανονισμό του Συμβουλίου. Ξεκινάμε με το άρθρο 4, παραγράφος 1, τροπολογία 45 του κυρίου Ζήλε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε τη 47 παρακαλώ, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, Ζήτω συγγνώμη, το ΕΛΚ κοίταζα. Ε, άρθρο 8, τροπολογία 2. Όχι, συγγνώμη, 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 49. Πρέπει να εγκριθεί. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 22 υπέρ, 19 κατά. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 9, 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία α υπέρ, Κατά. Α, συγγνώμη, χωριστή ψηφοφορία έχουμε εδώ. Πρώτο μέρος, μέχρι το rural. Ζητώ συγγνώμη από το ΕΛΚ. το πρώτο μέρος του συμβασμού υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος, με τη λέξη rural υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 55 όχι, 60. Η 55 καταπίπτει. 60 της κυρίας Τικάου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 11, 64, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 65, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 66, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 68, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 15, 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 έχει αποσυρθεί 74 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την 74 αρχή της πληροφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ποιος δεν ψήφισε, παρακαλώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 11, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 79 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 80 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 81. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 84 και 87 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Απορρίπτεται 86 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να πω κάτι, συνάδελφοι. Πολλέ από αυτέ τι ψηφοφορίε θα μπορούσαμε να τι έχουμε κάνει ε, μαζί, on block, αν κάποιο το είχε ζητήσει. Ε, τροπολογία 12 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ. Ε, ζητώ συγγνώμη, να ψηφίσουμε την 15, αρχή της ψηφοφορίας για την 15. Ψηφίσατε όλοι, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ. Ο κύριος Γκρός. Να ψηφίσουμε τις τροπολογίες του άρθρου 26 μαζί. 19 έως 106. την 19 ξεχωριστά. Να ψηφίσουμε πρώτα την 19 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95 με 106 μπορούμε να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι. 95 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 106 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με την ίδια πλειοψηφία απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Να την ελέγξουμε. 108. Αρχή της ψηφοφορίας για την 108. Ε, το ΕΛΚ δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει εκεί, τέλος πάντων, απορρίπτεται. 20 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, να, να ελέγξουμε την 115 αρχή της ψηφοφορίας. Everybody votes it. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 116 μαζί, μαζί με την 18 και 119. Υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε τις 116, 118 και 119, αρχή της ψηφοφορίας. Everybody voted. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Rejected. Απορρίπτεται. 23 those in favor. Those against. Abstain. Υπέρ, κατά, αποχές. Ε, απορρίπτεται. 117 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε την 117 αρχή της ψηφοφορίας. Ψήφισατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε, όχι απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 122 ε, υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 122, αρχή της ψηφοφορίας. How everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 124 παρακαλώ, αρχή της ψηφοφορίας. Τέσσερις σελίδες ακόμα συνάδελφοι. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε την 127 παρακαλώ, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 129 και 39 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 130 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 131 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 132, 134, 137 και 138. 40 και 46 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές. Να ελέγξουμε την 135 παρακαλώ, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 136. 43 και 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ τις τρεις αυτές τροπολογίες. Αρχή της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 139. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 141. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 140. Ε, να ελέγξω αν καταπίπτει ή όχι. Δεν καταπίπτει. τι ψηφοφορία έχουν ζητήσει η ECR. Το πρώτο μέρος ε, από το After the Midterm μέχρι το Basis. Το πρώτο μέρος λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε την 145 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να την ελέγξουμε. Εγκρίνεται. Τόσο λίγη σύγχυση υπάρχει. Ελέγχουμε την 26. Την 26 ελέγχουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλη η λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 152 και 153 ψηφίσω μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 και 157 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 και 159 μαζί υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 29 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 29. Αρχή της ψηφοφορίας για την 29. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 160, 162 και 170 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 172, 173, 174 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 175 και 176 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 178 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε παρακαλώ την 178 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι η λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε την 179. Νομίζω ότι η πλειοψηφία είναι η ίδια, αλλά να το ελέγξουμε. Αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Μετά έχουμε μαζί 48, 97, 100, 101, 102, ε, μέχρι την, την 171 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τα εκτιμώντας. 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε την 37 παρακαλώ, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 έχει αποσυρθεί. 42 της κυρίας Ενάλοβα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 42 αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, 180 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές να ελέγξουμε τις 43 παρακαλώ, αρχή της ψηφοφορίας. Everybody voted. Vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά αποχές 184 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τελική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε όλοι. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ, καμία κατά και 6 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Κράμερ για την έκθεση αυτή.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 So, Επομένως, ε, για έρευνα και ανάπτυξη έχουμε την επόμενη ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Ε, το Περιφερειακής Ανάπτυξης ξεκινούμε με τη τροπολογία ογκίας. Everybody ready to go on that? Είσαστε έτοιμοι να κάνουμε την ψηφοφορία. η τρίτη έκθεση του κ. Κράμερ, χειρουργίες. 50, πίνει υπέρ. Κατά, αποχές, 51 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται, 7 υπέρ. Εγκρίνεται, 52, Ταυτόση με την 7, 53, υπέρ, κατά yes, ε, εγκρίνεται 54 υπέρ κατά έλεγχος για την 54 ψηφίζουμε πέρας 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58, 59 και 60 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 9. Γιατί εγώ το είδα κάπου στο 3-2. Everybody voted. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 67. Κάντσον υπέρ κατά αποχές Έλεγχο για το 67. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Δεν κρίνεται. Και πάμε στο 70. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ένοχος 73. Ψηφίζουμε. Πέρας. απορρίπτονται. 75 πέρα. Αποχές. Και Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έχω στο 74 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται, Έλεγχος. Αλλά από ό,τι βλέπω το, το έλεγχο πρέπει να απέχει. 78 έλεγχος. Κύριο Σούγκερ και άλλοι δυο ψηφίσαν. Ε, πέρας. απορρίπτονται. 81. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Έλεγχος για το 81. Αυτή τη φορά νομίζω δεν σήκωσαν τα χέρια τους ή του ε, ομάδας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτονται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 87. Υπέρ. Υπέρ για το 87. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για το 87 ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 89. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 11. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 93. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 95 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεκατρία. Έχει αποσυρθεί 102. Πάμε στο 102, άλλες έχουν αποσυρθεί 102. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά χες εγκρίνεται 3 εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ Α, υπάρχει χωριστή ψηφορία εδώ όσον αφορά το αίτημα του ΕΛΚ. με ναι, ή χωρί την έκφραση rural, τη υπαίθρου, αγροτικό. Ναι ε, εγκρίνεται χωρίς με υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και άρα προστίθεται η λέξη rural συμβαστική γάμα C χωστή ψηφοφορία από το ECR όλο το κείμενο μέχρι εκεί που λέει υπάρχουσες υποδομές βρε, βρέχει χρόνια υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, 116. Όχι, 117 λέει ο 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Α, απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική δέλτα χωρική ψηφοφορία πάλι για το rural το πρώτο τμήμα με το rural μα γιατί, γιατί έχετε κολλήσει με το rural ε, αυτή ποιο είναι υπέρ του για το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συνεχίζει και είναι δημοφιλή η λέξη rural από ό,τι βλέπουμε. Τώρα πάμε στο 25 με την προφορική τροπολογία. Αντιγράφουμε για να υποκαθιστούμε εδώ τη, τη λέξη basic με τη λέξη fundamental βασικός με θεμελιώδης. Οπότε θα γίνει αυτή η αλλαγή, προτείνεται, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές και εγκρίνεται συμβιβαστική, ε, ε, να από εδώ πέρα το rural δεν ξαναφύτρωσε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 132. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος για το 132. Ψηφίζουν. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται 131 κατά αποχές εγκρίνεται. 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 έλεγχος 138 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται 6 προφορική. Ε, εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία, ελπίζω συμφωνείτε. Επίσης έχουμε και την προσθήκη που έχει στηθεί από το ΕΛΚ. Επομένως θα κάνουμε την προφορική τροπολογία πρώτα και μετά την προσθήκη. Για την προφορική τροπολογία υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τώρα η προσθήκη, είναι υπέρ είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τι βασανιστήριο. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 140. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 145 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για το 145 ψηφίζουμε. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Εγκρίνεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, έλεγχος 147. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι.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 απορρίπτεται 151. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 152. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153. Υπέρ. Κατά, Κατά έλεγχος για το 153. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 156 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές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 εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ψηφίζουμε πέρας απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 Ψήφισαμε μόνο το πρώτο τμήμα, το δεύτερο έχει αποσυρθεί. Το πρώτο. Περιβάλλον. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα κάνουμε έλεγχο για το 6 ψηφίζουμε ψήφισαν όλοι πέρας και εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στο παράδειγμα. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 157 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, δεν έχει αποσυρθεί, 164 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος. 164. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Έλεγχος. 165. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 66. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Το 35 υπέρ 0 κατά 2 αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τώρα στην επόμενη. Which one's this one now? This one. Starts with amendment eight. Yes. Right. The next one is. Η επόμενη γνωμοδότηση αφορά το Ταμείο Συνοχής. Το άρθρο 2 ξεκινάει με την τροπολογία 8. I'll be waking up in the middle of the night going for against the opposition. Τροπολογία 8. Είμαστε έτοιμοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Έτσι λοιπόν περνάμε στην 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 37 ξεκινά η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται 3 Άρθρο 3, η 11 έχει αποσυρθεί, συμβιβαστική ήττα με χωριστή ψηφοφορία. Εδώ έχουμε τον φίλο το η λέξη rural, ξανά το πρώτο μέρος χωρίς, ε, υπερκατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο μέρος προσθήκη της λέξης rural, υπερκατά κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεκαπέντε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική G το rural πάλι πρώτο κομμάτι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος, προσθήκη της λέξης rural, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παίρναμε τώρα στη συμβιβαστική γιώτα. Δεν έχουμε το rural εδώ, συμβιβαστική γιώτα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική J, πρώτο μέρος. Με το Interoperable Transport and Mobility διαλειτουργικές μεταφορές και κινητικότητα. Τέσσερα μέρη έχει αυτή το, η συμβιβαστική. Τέσσερα μέρη. Έχουμε, πώς γίνεται να έχουμε μια συμβιβαστική που την οποία χωρίζουμε σε τέσσερα μέρη δεν το καταλαβαίνω. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται δεύτερο μέρος. Καρπούλινγκ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται τρίτο μέρος Sustainable Urban Mobility, υπέρ κατά, αποχές. Ελέγχουμε το τρίτο μέρος, ξεκινάει ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τέταρτο μέρος υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε το τέταρτο μέρος. Ξεκινάει η ψηφοφορία στο τέταρτο, για το τέταρτο μέρος. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Το τέταρτο αυτό μέρος απορρίπτεται συμβιβαστική κάπα τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 58 ξεκινάει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι κλείνει Απορρίπτεται. 59 Σνάλοβα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρθρο 4 προφορική τροπολογία L λάμδα όλοι ικανοποιημένοι και μετά έχουμε την προσθήκη του ΕΛΚ. Πρώτα την προφορική τροπολογία δεν έχει αντίρρηση υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα η προσθήκη του ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 61 παρακαλώ ξεκινάει η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ καταπίπτει 63 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές να ελεγξούμε το 2 ξεκινάει η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι κλείνει απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 30 ε, άρχιτη ψηφοφορία ψήφισαν όλοι κλείνει ψηφοφορία εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 67 και 68 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 αποσύρεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 72 ξεκινάει η ψηφοφορία Ψήφισαν άπαντε, κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 23 ε, του εισηγητού υπέρ κατά. Από 23 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 73. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Κλείνει ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται τελική ψηφοφορία. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ξεκινάει ανάπαντος. Κλείνει ψηφοφορία. 34 υπέρ. 4 αποχές. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στο Μάκη και για τις τρεις νομοδοτήσεις. Και συγχαρητήρια στα μέλη για τις μαραθώνιες ικανότητές τους να επιβιώνουν μετά από μια τέτοια μακρόχρονη ψηφοφορία. Yeah, but I'll need uh, Dominic to take over at 11.15 because I've got to go. Dominic, could you take over at 11.15? Shall we bring the minister Take over, yeah. Yes.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 Okay, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας ενημερώσω ότι εγώ θα εγκαταλείψω την Προεδρία στις 11 και 4 για να παραστώ στη συνεδρίαση με τον Πρόεδρο για το Πολιτές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και ο Ντομινίκ θα αναλάβει ως Πρόεδρος για τη συνεδρίαση με τον Υπουργό. Ζητούμε συγγνώμη γιατί η καθυστέρηση, κύριε Υπουργέ, ήταν επειδή οι ψηφοφόροι ε, διήρκεσαν πολύ, αλλά καθώς ο συναδελφός ο κύριος Σόν δεν θα παρευρίσκεται μαζί μας, ε, δεν είμαστε τόσο πιεσμένοι από το χρόνο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τον Δανό Υπουργό Μεταφορών, Henrik Dam Christensen. Ήρθε εδώ για να μας ε, παρουσιάσει μια έκθεση για την Δανική Προεδρία. Καλώς ήρθατε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, και έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ευρωβουλευτές ε, δεν πρέπει να ζητάνε συγγνώμη για να κάνουν τη δουλειά τους. Ε, η ψηφοφορία είναι πολύ σημαντικό μέρος της δουλειάς των ευρωβουλευτών. Μην ζητάτε λοιπόν συγγνώμη γι' αυτό. Και Πράγματι ο συνάδελφός μου ο Λεσόν δεν ε, μπορεί να πάρει το λόγο, δεν μπορεί να παρευρεθεί και να μιλήσει για τα ε, ναυτιλιακά θέματα. Γι' αυτό ε, υποσχέθηκα να μιλήσω και για τα θέματα αυτά. Δεν είμαι ειδικό, θα προσπαθήσω να απαντήσω, αλλά κατά τα άλλα σας πω ότι μπορούμε να σας απαντήσουμε και γραπτώς σε ενδεχόμενες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να επανέλθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Τραν και να ε, σας πω λίγα λόγια για το περασμένο εξάμεινο της Προεδρίας μας. Ε, θα θυμάστε ότι αναλάβαμε τη σκητάλη από την Πολωνία και σε λίγο θα είναι η σειρά της Κύπρου. Θα ήθελα να πω ότι περάσαμε πολύ ενδιαφέροντες καιρούς, ε, πολύ σκληρή δουλειά έκαναν όλοι όσοι συμμετείχαν και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για τη στενή συνεργασία που είχαμε με το Κοινοβούλιο. Ε, πολύ σκληρή δουλειά κάναμε σε συνεργασία μαζί σας και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτήν. Η Δανέζικη Προεδρία ε, επικεντρώθηκε στις, ε, στην πράσινη ανάπτυξη ως ε, δρόμο εξόδου από την κρίση. Όλοι ξέρουμε ότι η υποδομή και ο αποτελεσματικός τομέας μεταφορών αποτελούν σημαντική κινητήρια ε, δύναμη για την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Χαίρομαι επίσης που καταφέραμε να προωθήσουμε μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Ε, θα ήθελα να επικεντρωθώ ιδιαίτερα στα εξή δύο από τις προτάσεις στο πακέτο αεροδρομίων, η πρόταση ε, για τις υπηρεσίες εδάφους ε, και για την ε, μείωση του θορύβου στα αεροδρόμια της Ευρώπης είναι πολύ σημαντικέ. Επίσης είχαμε την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Έχουμε την διευκόλυνση Connecting Europe ενώνοντας την Ευρώπη. Και έχουμε και το θέμα του συστήματος πλοήγησης Γαλιλαίου και

Ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί πολύ το Κοινοβούλιο είναι η αναθεώρηση του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων. Στον τομέα των αεροδρομίων έχουμε κάνει, έχουμε ε, κάνει σημαντικές πρόοδους και η πρόταση για τις υπηρεσίες εδάφους και η πρόταση για την μείωση της ε, ηχοστάθμης ε, είναι σημαντικά θέματα. Τα αεροδρόμια είναι σημαντικός τρόπος να ενωθεί η Ευρώπη και τα δύο πακέτα αυτά βελτιώνουν τις υπηρεσίες και το δυναμικό στα αεροδρόμια της Ευρώπης. Οι εργασίες για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών για τα διευρωπαϊκά δίκτυα αποτέλεσε προτεραιότητα και κατά την ε, Πολωνική και κατά την Δανέζικη Προεδρία και υπήρχε ισχυρή βούληση να προωθηθεί η πρόταση αυτή όσο γίνεται περισσότερο εντύπωση μου είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη ήθελαν να συμβάλλουν ώστε να έχουμε καλό πλαίσιο για τις επενδύσεις του μέλλοντος να μπορέσουμε στο, στα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε ένα συνεκτικό σύστημα μεταφορών που θα διευκολύνει τις συνοριακές μετακινήσεις στην ε, Ευρώπη. Η, μια καλή υποδομή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και γι' αυτό η πρόταση αυτή έχει ε, σημαντικό δυναμικό για την οικονομία της Ευρώπης και γι' αυτό χαίρομαι που ήδη στο Συμβούλιο της 22ης Μαρτίου επιτεύχθη η συμφωνία. Θα πρέπει να δούμε την πρόταση αυτή μαζί με τα κριτήρια για την ε, κατανομή των ε, διευρωπαϊκών ε, δικτύων. Χαίρομαι που η βούληση του Συμβουλίου συνεχίστηκε και στις 7 Ιουνίου επιτεύχθη συμφωνία σχετικά με την δημιουργία της διευκόλυνσης Connecting Europe νέες κατευθυντήρες γραμμέ για τα διευρωπαϊκά δίκτυα από το CEF θα είναι πολύ σημαντικά ώστε να διασφαλίσουν ε, σημαντικά διασυνοριακά έργα τα οποία κατά τα άλλα δεν, ήταν, δεν θα ήταν δυνατά να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν και έτσι να κλείσουμε τα κενά στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Έχουμε δύο δύσκολα θέματα για επενδύσεις ε, στα κράτη-μέλη που ταυτόχρονα καθορίζουν ε, οι ε, χρηματοδότηση μπορούν να λάβουν τα κράτη-μέλη στο διάστημα 2014-2020 για σημαντικά θέματα υποδομών. Στο Συμβούλιο της 7ης Ιουνίου επιτεύχθη συμφωνία σχετικά με την ε, πρόταση για δημιουργία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Δορυφόρων Γαλιλαίο. Έχουμε κάνει λοιπόν ένα σημαντικό βήμα ε, για την πλήρη λειτουργία του Γαλιλαίου το έτος 2020. Όσον αφορά την αναθεώρηση του πρώτου πακέτου σιδηροδρόμων, στόχος μας ήταν να πετύχουμε λύση στο, κατά τη δεύτερη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο για να επιτευχθεί συμφωνία στην πρόταση αυτή. Ε, με χαρά μπορώ να σα πω ότι σήμερα στην Κορεπέρη υπήρχε υποστήριξη προ την ε, πρόταση τη Κομισιόν. Ε, βρίσκω θετικό το ότι επιτεύχθη η συμφωνία στην πρόταση αυτή που ως γνωστόν είναι σημαντικό κομμάτι για την ε, ε, ε, για την σωστή λειτουργία των συνδεδεμένων στην Ευρώπη. Θα ήθελα να συγχαρώ την, ε, το Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα των ε, διαπραγματεύσεων. Επίσης έχουμε την πρόταση για συστήματα ελέγχου στον τομέα των μεταφορών για να βελτιωθεί ο έλεγχος και να μειωθεί το οικονομικό άχθος για τις εταιρείε μεταφορών. Ε, κατά τα άλλα, έχουμε επικεντρωθεί σε τρία θέματα. Στις 22 Μαρτίου συζητήσαμε το θέμα της ασφαλείας στα αεροδρόμια, διότι μας απασχολεί το ότι οι κανόνες ασφαλείας γίνονται όλο και πιο πολύπλοκοι για τις ε, ε, αεροπορικές εταιρείε και τους επιβάτες χωρίς να επιφέρουν θέμενη αξία. Οι κανόνες θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική βάση. Σημαντικό είναι οι επιβάτες να γνωρίζουν ότι είναι ε, ξεκούραστοι και ικανοί να ε, διεξάγουν την ε, πτήση, οι πιλότοι και τα πληρώματα. σημαντικό είναι, σημαντική είναι επίσης η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη στις 17 Απριλίου του 2012 ε, σχετικά με το σύστημα WLTS όπου μπορέσαμε να να ε, ανταλλάξουμε εμπειρίες σχετικά με το σύστημα EMTS στην Ευρώπη. Ε, και στις 7 Μαΐου είχαμε διάσκεψη για σημαντικά έργα υποδομών και είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στα θέματα αυτά στους δύσκολους αυτούς καιρούς. Και τέλος, ε, στις 27 Ιουνίου έχουμε μια ε, διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την ε, οδική ασφάλεια στην Κοπεχάγη. Σας ε, παρουσιάσω τώρα τα ναυτιλιακά θέματα, διότι ο συνάδελφός μου ο Λεσόν δεν μπορεί να είναι παρόν, αλλά με παρακάλεσε να σας παρουσιάσω τα εξής. Ε, καταρχήν, μου ζήτησε να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας ε, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Brian Simpson για την στενή και επικοδομητική συνεργασία κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας. Η Δανέζικη Προεδρία κυρίως έχει επικεντρωθεί στις τροποποιήσεις ε, του της σύμβασης STCW, ε, αναθεώρηση του κανονισμού ΕΜΣΑ, ε, τον κανονισμό για τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους και την Διεθνή Σύμβαση για την Ναυτική Εργασία. Όσον αφορά την οδηγία STCW, ελπίζουμε σήμερα ότι στον τριμερή διάλογο ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την ε, συμφωνία αυτή. Ε, βελτιώνεται η εκπαίδευση των ε, ναυτικών και με πιο αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις περιόδους ανάπαυσης και την κατανάλωση αλκοόλ. Επικεντρωνόμαστε και στις τις προσπάθειες κατά της πειρατείας. Ε, όσον αφορά τον κανονισμό ΕΜΣΑ, ε, προσπαθήσαμε να επιτύχουμε συμφωνία με το Κοινοβούλιο με ισορροπημένο τρόπο και γι' αυτό με μεγάλη χαρά μας ε, στις 12 Απριλίου 2012 διαπιστώσαμε ότι καταλήξαμε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης έχουμε την συμφωνία για τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους για να μπορέσουμε να έχουμε πιο με την συμφωνία αυτή είχαμε το πρώτο αποτέλεσμα για την Δανέζικη Προεδρία στα θέματα ναυτιλίας τον Απρίλιο. Ο κανονισμός ε, αυτός ε, ε, μαζεύει όλες τις τροποποίησεις που έχουν γίνει από το 2002 και έτσι υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τους κοινοτικούς κανόνες. Σημαντικό θέμα που μας έχει απασχολήσει κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας είναι το θέμα της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για την ναυτική εργασία. Θα ήθελα σύντομα να αναφερθώ στην πειρατεία που είναι μια από τις σημαντικότερες ε, κατά τη ναυτιλία σήμερα. Γι' αυτό με μεγάλη μα χαρά μπορέσαμε να οργανώσουμε την τρίτη διάσκεψη για την πειρατεία τον Μάρτιο του 2012. Η διάσκεψη αυτή έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε ε, στην ε, διεθνή προσπάθεια κατά πολέμηση τη πειρατεία. Και ο συνάδελφό μου, ο Λεσόν, καταλήγει ότι ε, και στον αγώνα κατά τη πειρατεία έχουμε σημειώσει βήματα πρόοδου. Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να πω ως ε, αναφορά από την Δανέζικη Προεδρία. Να σας ευχαριστήσω για την στενή συνεργασία που είχαμε ε, με την Επιτροπή Τραν. Ε, προσωπικά την εκτίμησα ιδιαίτερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτα πρώτα να μιλήσουν οι συντονιστές. Κύριος Γκρός πρώτα για το ΕΛΚ. Αλλά πρώτα-πρώτα παρακαλώ να κάνουμε την ε, εναλλαγή εδώ στην Προεδρία ε, γιατί πρέπει να πάω στην υποχρέωση που σας είπα, στην συνάντηση εκείνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Συμβουλίου για την ε, δουλειά της. Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να βρίσκονται λύσεις και συμβιβασμοί με τις οποίες μάλιστα δεν συμφωνούν πάντα όλοι. Σύντομα, ένα από τα σημαντικότερα θέματα ε, παραμένει για μας το θέμα των διευρωπαϊκών δικτύων και του CEF. Ελπίζουμε το Συμβούλιο και οι εκπρόσωποι των μεταφορών στο Συμβούλιο να ε, συνεχίσουν να συμφωνούν ε, στο θέμα αυτό και είπατε και το επαναλαμβάνουμε και εμείς στο Κοινοβούλιο, το θέμα δεν είναι πού θα βρούμε χρήματα αύριο. Θα πρέπει... Ε, το θέμα δεν είναι μόνο να μειώσουμε τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε και κάποια έργα. Στο θέμα αυτό είναι σημαντικό να, έχουμε, να ενεργούμε με αποφασιστικότητα και Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε τις ε, υποδομές μεταφορών ε, επιπλέον δαπάνη στα κράτη-μέλη, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση. Σήμερα δεν θα εμβαθύνουμε περαιτέρω στο θέμα αυτό. Ελπίζουμε όμως ότι εσείς με τις εμπειρίες της Προεδρίας σας θα συνεχίσετε να βρίσκεστε στο πλευρό μας ε, όταν ε, θα ακολουθήσουμε τη γραμμή αυτή και όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και όσον αφορά την ε, διευκόλυνση ενώνοντα την Ευρώπη. Όσον αφορά την αναδιατύπωση, το, αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό σήμερα. Θέλουμε ισχυρό ρυθμιστικό φορέα στα κράτη-μέλη, ε, ενδεχομένως ε, με ένα δίκτυο. Αυτό είναι σημαντικό σημείο πρόοδου. και Σημαντικό είναι να έχουμε και έναν ε, σωστό διαμεσολαβητή που να ελέγχει τον ανταγωνισμό στα κράτη-μέλη. Ελπίζουμε ότι Πολωνοί συνάδελφοι μπορούν να συμφωνήσουν. Αλλά ξέρετε ότι ακόμα και ο καλύτερο συμβιβασμό μπορεί την τελευταία στιγμή να βελτιωθεί. Δεν έχουμε καταλήψει λοιπόν κάθε ελπίδα. Θα ήθελα επίσης ε, να σας πω ότι θέλουμε να αδράξουμε την ευκαιρία ώστε να επιφέρουμε προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και για τους οδηγούς. Θέλουμε λοιπόν να σημειώσουμε βήματα πρόοδου ώστε οι οδικές μεταφορές ε, να μην αποτελεί ε, χώρο για ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Από και από οικονομικής πλευράς είναι σημαντικές οι κοινωνικές πτυχές, ε, διότι ε, παίζουν σημαντικό ε, οικονομικό ρόλο οι ε, μεταφορές. Στον συνάδελφο Κράμερ θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν διστάμενες απόψεις για διάφορα θέματα και εγώ μιλώντας τελείως προσωπικά Σημερίζομαι την ερμηνεία της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει, ε, να πω ότι, θα πρέπει να είμαι δίκαιος και να πω ότι ε, τη θέση αυτή δεν την ε, συμμερίζονται και άλλοι, αλλά είναι ένας διάλογος που θα πρέπει να διεξάγει το Κοινοβούλιο με την Κομισιόν. Είναι σημαντικό οι πολίτες να βλέπουν και τη διαδικασία. Διότι αν σήμερα μια ερμηνεία ε, ε, ε, ακολουθήσει μια κατεύθυνση και σε δύο χρόνια ακολουθήσουμε μια άλλη ερμηνεία, τότε δημιουργούμε ανασφάλεια στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις λένε μπορώ να αγοράσω σήμερα τέτοια φορτηγά, αν σε τρία χρόνια θα έχουμε μια τρίτη ερμηνεία και μου πείτε ότι είναι παράνομα τα οχήματα αυτά. Αυτό είναι το δύσκολο στην κατάσταση αυτή. Χρειάζεται, ε, απαιτείται κατά τη γνώμη μου πολύ περισσότερη νομική ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε την ε, διαδικασία από το περιεχόμενο. Όσον αφορά τον ε, τομέα των αερομεταφορών, έχει φτάσει το θέμα στο Συμβούλιο. Εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε κάποιες πτυχές. Υπάρχουν κάποιες πτυχέ οι οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη συζήτηση. Θα θέλω να αναφερθώ στην ηχοστάθμη. Και πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ε, μια ε, πιο ε, καλή εφαρμογή της επικουρικότητας και εντός της Ευρώπης και εκτός. Όσον αφορά τα σλότς, θα πρέπει να το θέμα είναι κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια βελτίωση και όσον αφορά τις υπηρεσίες εδάφους, χρειαζόμαστε σωστές ε, συνθήκες εργασίας σε έναν πολύ δύσκολο τομέα. Ερώτησή μου είναι... Δεν ξέρω γιατί, αλλά όσον αφορά τον ε, ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό έχουν γίνει πολύ λίγα. Ε, πολύ λίγα πράγματα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να γίνει κάτι. Είναι απόλυτα δικαιολογημένες οι προσδοκίες αυτές. Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες και βρίσκω ότι είναι σημαντικό όταν λαμβάνουμε από κοινού ε, μία ε, απόφαση θα πρέπει να γίνεται σεβαστή αυτή. Πριν ε, δύο-τρία χρόνια έχουμε λάβει μια απόφαση, ε, αλλά τώρα αρνούμαστε να την εφαρμόσουμε. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό και δεν ε, κατηγορώ εσάς, αλλά ελπίζω η επόμενη Προεδρία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Πιστεύω όμως ότι απαιτείται κάθε Προεδρία να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ακούσω την θέση σας για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχετε κάνει σε αυτούς τους όχι πολύ εύκολους καιρούς. Ευχαριστώ κύριε Γκρός, ο κύριος Χαντραούι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τη Δανική Προεδρία για τα όσα έχει πράξει μέχρι σήμερα. Ήσασταν πάρα πολύ δραστήριοι και πολύ παραγωγικοί. Κάναμε σημαντικά βήματα προς τα εμπρός. Συγχαρητήρια λοιπόν. Αυτό αποδεικνύει για άλλα μια φορά το γεγονό ότι οι μικρότερε χώρε ορισμένε φορέ ε, στην πραγματικότητα μπορούν να επιτύχουν πολλά με την Προεδρία του Συμβουλίου από τι μεγαλύτερε χώρε. Έχω μερικέ παρατηρήσει να κάνω. Αν και στα περισσότερα αναφέρθηκε ο προηγούμενο συνάδελφο, όσον αφορά τι μελλοντικέ μεταφορέ πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το CF. Αυτό ίσως είναι το σημείο το πιο σημαντικό. Έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός και θα πρέπει και εμείς, όπως είπε ο συνάδελφος, με τον οποίο συμφωνώ, όπως είπε ότι τα κονδύλια του συνδέοντας την Ευρώπη, του μηχανισμού συνδέοντας την Ευρώπη αποτελούν βασικό κομμάτι, διότι αλλιώς το όλο θέμα είναι κενό και μας ανησυχεί ω κοινοβούλιο αυτές τις τυχόν θέσεις που ορισμένοι συνάδελφοι από εσάς από τον προπολογισμό ενδεχομένως μπορούν να υιοθετήσουν. Και η Δανία προτείνει το γενικός προπολογισμός ε, να μην υπάρχει μεγάλο χάσμα. Υπάρχει φόβος ότι αυτό το επενδυτικό ταμείο θα αποτελέσει το θύμα της συζήτησης. Ελπίζω ωστόσο ότι στους επόμενους μήνες ε, θα κάνετε ό,τι μπορείτε όσον αφορά τις αερομεταφορές και τα αεροδρόμια. Το μελετάμε Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της άσκησης, θα το σκεφτούμε και θα σας ενημερώσουμε. Επίσης μου φαίνεται ότι είναι σημαντικό ε, να δούμε τα αποτελέσματα της αναδιατύπωσης μετά από τους συμβιβασμούς του τριμερούς διαλόγου της περασμένης εβδομάδας. Ε, πρόκειται για μια επιτυχή ιστορία, αναμφίβολα. Ίσως ορισμένοι δεν είναι ευχαριστημένοι απολύτω με του συμβιβασμού, ωστόσο προχωράμε υποστηρίζοντας τη διαφάνεια, διότι το σιδηροδρομικό σύστημα είναι σημαντικό και το Κοινοβούλιο ισχυρίζεται ότι θέλει να ενισχύσει τη θέση του νομοθέτη. Και μετά την περασμένη εβδομάδα συζητήσαμε για την απελευθέρωση την αποδεσμοποίηση μεταξύ των διαχειριστών των υποδομών, των φορέων ε, είναι σημεία που απασχολούν όχι μόνο το Κοινοβούλιο. Θεωρώ ωστόσο ότι η θέση όπως έχει μέχρι σήμερα αποτελεί βήμα προς τα μπρος ένα άλλο σημείο αφορά την ενίσχυση του ευρωπαϊκού, ε, της Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Υπηρεσίας. Ε, σύμφωνα με τις συζητήσεις θέλουν να δημιουργηθούν νέα μέτρα, ενίσχυση των μέτρων και μετά άλλα δύο σημεία που μου φαίνονται σημαντικά όσον αφορά το Single Sky δεν έχουν γίνει και πολλά. Η προθεσμία είναι Δεκέμβριο του 2012, όχι... Είναι δίπλα μας και ε, ελπίζω ότι οι Κύπροι συνάδελφοι θα διατηρήσουν θα, θα επιταχύνουν ώστε όλα τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να καταλήξουν σε κάτι μέχρι τα του 2012 ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τα ε, επιχειρησιακά σημεία. Ένα άλλο σημείο όσον αφορά τα μεγάλα φορτηγά, τα μεγατήρ. Υπάρχουν διάφορες θέσεις ε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το θέμα για αυτούς τους κύκλοπες των δρόμων το σημαντικότερο είναι να δούμε κατά πόσο η στρατηγική που αφορά αυτά τα οχήματα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια. Αυτό ίσως να χρειαστεί να αλλάξουν οι νομοθεσίες και αυτό βάσει δημοκρατικών συζητήσεων το Ευρωκοινοβούλιο ακούτε επιχείρηματα υπέρ και κατά. Εσείς γνωρίζετε τις δικές μας απόψεις, ξέρετε τι θεωρούμε ότι δεν πάει καλά, αλλά είναι λίγο περίεργο που αυτές οι ρυθμίσεις ξαφνικά ερμηνεύονται διαφορετικά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα της Κομισιόν μας ανακοινώνουν μάλιστα ότι σε μερικούς μένες θα γίνει μια τροποποίηση που θα μας παρουσιάσουν, ίσως να έχουμε κάτι καινούριο. Συνοπτικά αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν ορισμένα σημεία σύγχυσης ε, για το μέλλον. Ε, συγχαρητήρια για τη Δανική Προεδρία φυσικά. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας. Ελπίζουμε να σας ξαναδούμε σύντομα και θα αξιοποιήσουμε την οριμότητα και την εμπειρία και ελπίζουμε ότι ως μελλοντικό μέλος του, ε, του Συμβουλίου θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εμπειρία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μας ε, παρουσιάσατε τα αποτελέσματα της εργασίας σας ε, και όπως είπατε κατά τη διάρκεια της Δανείσκης Προεδρίας ε, έχει σημειωθεί η πρόοδος σε πολλά θέματα. Ε, εμείς το Κοινοβούλιο Όλε ε, οι πολιτικέ ομάδε, μάλιστα, που διότι ξέρετε ότι δεν συμφωνούμε πάντα, στηρίζουμε το θέμα ε, των διευρωπαϊκών δικτύων. Και είπατε ότι στο Συμβούλιο προσπαθήσατε να δημιουργήσετε ένα ε, καλό χρηματοδοτικό πλαίσιο. Νομίζω ότι έτσι το είπατε. Ξέρουμε όμω ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποιε χώρε που πιστεύουν ότι τα, το, το χρηματικό ποσό των 50 δισεκατομμυρίων είναι υπερβολικά μεγάλο για το επόμενο χρονικό διάστημα, ότι προχωράμε πολύ γρήγορα. και ελπίζω ε, ε, εσείς ε, να μπορείτε να πείσετε τους συναδέλφους σας ότι είναι κάτι που θα ωφελήσει το σύνολο της Ευρώπης αν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τα έργα αυτά. Επίσης, όσον αφορά τα ομόλογα μεγάλων έργων, εάν μπορέσουμε να τα προωθήσουμε, αυτά θα είναι καλό, διότι νομίζω ότι αν μπορέσουμε να δείξουμε ότι με ε, τα 230 εκατομμύρια μέχρι το τέλος του 2013 θα μπορέσουμε να πετύχουμε ε, ένα αποτέλεσμα μόχλευσης. Ε, αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία και αν μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο για τα 31,7 εκατομμύρια στον τομέα των μεταφορών, πιστεύω ότι αυτό θα προωθήσει την Ευρώπη. Γι' αυτό το πιο σημαντικό από όλα είναι να στηρίξουμε αυτή την πρόταση της Κομισιόν, διότι νομίζω ότι ε, θα ωφελήσει όλους μας εδώ στην Ευρώπη. Επίσης ε, αναφερθήκατε στην ψηφιακή τεχνολογία. Θα πρέπει να ε, είναι μικρότερο το άχθος για τις επιχειρήσεις και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε για την Κομισιόν. Από την ομάδα στο Ήπερι και από την Κομισιόν ε, υπεγράφει μια πρόταση, από, ε, ε, μια πρόταση σχετικά με την μείωση του αχθούς Υπάρχουν διστάμενες απόψεις για την πρόταση αυτή, αλλά υπήρχε συνένεση ότι θα ήταν ε, λογικό τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να τις απαλλάξουμε από το υπερβολικό διοικητικό κόστος. Περιμένω λοιπόν να δω τι θα γίνει με αυτούς τους ψηφιακούς ταχυγράφους. Επίσης, ε, κάποια θέματα δεν θα μπορέσουν να κλείσουν κατά διάρκεια της Προεδρίας σας. Ε, όσον αφορά την, ε, τις αερομεταφορές, για μένα σημαντικό είναι να αναφέρω τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Είναι ένα θέμα το, οποίο φαίνεται να αποτυγχάνει. Εσείς ως ε, Δανός υπουργό μπορεί να μην μπορέσετε να κάνετε πολλά για το θέμα αυτό. Ε, θα πρέπει και η Γερμανία και η Γαλλία να ε, κάνουν επιτέλους κάτι. Πάντως, Εμά μα ενδιαφέρει να τονίσουμε ότι χρειαζόμαστε βελτίωση στο θέμα αυτό. Όσον αφορά την αναδιατύπωση για του σιδηροδρόμου, ναι, μα αρέσει το θέμα των ρυθμιστικών αρχών. Ε, πιστεύουμε επίσης ότι είναι σωστή, σωστό το να γίνει η διάκριση, ε, να γίνει ο διαχωρισμός ε, των λειτουργών των δικτύων. Θα κλείσω το θέμα αυτό διότι δεν θέλω να μακρηγορήσω. Όσον αφορά τα μεγάλα φορτηγά, τα οποία έχουν διάφορες ονομασίες και Ecoliner τα ονομάζουν, δεν είναι ότι είναι λάθος το όνομα αυτό, αλλά υπάρχουν στάμενες απόψεις. Εγώ προέρχομαι από την κάτω Σαξονία και διαπιστώθηκε εκεί ότι είναι η οικονομική και η οικονομική η χρήση των φορτηγών αυτών σε, κάποια, σε κάποιες ε, περιφέρειες. Και ακριβώς ε, γι' αυτό με στεναχωρεί το ότι με τη συζήτηση αυτή και με την επιστολή του Επιτρόπου υπάρχει νομική ανασφάλεια και οι επιχειρήσεις ε, δεν γνωρίζουν ε, πώς έχει η κατάσταση, δεν έχει ξεκαθαριστεί αν μπορούν να περνούν τα σύνορα από τις κάτω χώρες ε, στην κατοσαξονία, τι γίνεται με τη Δανία, τη Σουηδία. Χρειαζόμαστε εδώ περισσότερε πληροφορίε. Ε, νομίζω ότι δεν μπορείτε κι εσεί να κάνετε πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, αλλά θα προσπαθήσω με, το, με την Κομισιόν ε, και το Κοινοβούλιο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε νομική βεβαιότητα. Όσον αφορά τα θαλάσσια θέματα, εσείς πήρατε το λόγο εκ μέρους του Συναδέρφους σας. Ε, Παρ' όλα αυτά τα δεξαμενόπλια διπλού του πιστεύω ότι είναι πολύ καλό πράγμα. Ε, είχαμε κάποιες, κάποια ατυχήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ καλό το ότι έχουμε προχωρήσει στο θέμα, στο θέμα αυτό. Επίση, η βελτίωση των συνθήκων ε, των ναυτικών καθώ και το θέμα Τη ε, ναυτική εργασία, ε, διότι θέλουμε ε, να έχουμε εργαζόμενου στον τομέα αυτό, αλλά αν δεν είναι ολκυστικό ο τομέας δεν θα έχουμε το απαραίτητο δυναμικό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή και τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Όσον αφορά την πειρατεία, έγινε μια διάσκεψη και σε συνεργασία με την Κομισιόν, την βρήκα καλή, μπόρεσα να συμμετάσχω εν μέρη. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα τη καταπολέμηση τη πειρατεία. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε και τις αιτίες. Δεν είναι μόνο θέμα μεταφορών, είναι και θέμα Εξωτερική εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής ε, και πολιτική ασφαλείας. Αλλά ε, είναι κάτι που επηρεάζει ιδιαίτερα τον τομέα των μεταφορών και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι θετικό ε, το ότι κάνατε κάποια πράγματα κατά τη διάρκεια τη Προεδρίας σα και ότι οι Δανείοι είπαν ότι ναι, είμαστε ειρηνικός λαός, αλλά ε, και εμείς ε, έχουμε ε, καταβάλει προσπάθειες ώστε να προστατεύουμε το, τα πληρώματά μας. Ε, όσον αφορά την ε, ΕΜΣΑ, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό επειδή θα έχουμε και τη συζήτηση για το προπολογισμό, ότι θα θέλαμε να έχουμε μια επιπλέον αρμοδιότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι σημαντικό για μας ε, να ε, πρικοδοτηθεί σωστά και η ΕΜΣΑ. Και τέλος έχω μία ερώτηση για έναν τομέα στον οποίο δεν αναφερθήκατε. Δεν ξέρω αν είναι ε, υπεύθυνο, αν είναι αρμόδιος ο συναδελφός σας, έχει να κάνει με την, ενιαία θαλάσσια, την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Το Συμβούλιο μας είπε ότι φέτος και του χρόνου 50 ε, εκατομμύρια ευρώ ε, θα διατεθούν και άκουσα ότι το Συμβούλιο θέλει να μειώσει τη χρηματοδότηση. Ε, ισχύει αυτό, γνωρίζετε κάτι για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν με το στον κύριο Κράμερ. Να ευχαριστήσω και εγώ ε, τον Δανό Προεδρεύοντα. Είχαμε στενή συνεργασία, στενές επαφέ ε, παρότι δεν συμφωνούσαμε πάντα, αλλά πήρατε πολύ σε σοβαρά το έργο σας, ε, ε, εργαστήκατε σκληρά. Όσον αφορά την αναδιατύπωση μπορεί να μην υπήρχαν πολλά προβλήματα. Σε άλλα θέματα όμως μπορεί να είχαμε ε, διαφωνίες ε, σε κάποια ε, θέματα. Ακούσαμε δηλώσεις λίγο περίεργε, όχι από εσά, αλλά από άλλους προσώπου της Δανία. Ε, όσον αφορά τα σημαντικά θέματα, έχουμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα και ε, τα σχετικά θέματα. Από το Συμβούλιο και το και την Κομισιόν. Ε, θα ήθελα μια ανάλυση. Εδώ και 30 χρόνια ε, θέλαμε να κάνουμε ε, μια σχετική ανάλυση και ε, τα τελευταία 30 χρόνια μάλλον είχαμε περισσότερα χρήματα από θα έχουμε τα επόμενα 30. 20 δισεκατομμύρια ήθελαν το, η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο ενώ τελικά καταλήξαμε σε 8 λόγω του Συμβουλίου τα προβλήματα φαίνεται να υπάρχουν πάντα εκεί που είναι τα σύνορα και εγώ θα ήθελα λοιπόν μια ανάλυση της ε, συνολικής πολιτικής. Ε, ποντάρουμε υπερβολικά πολλά ε, στα μεγάλα έργα και οι Πολωνοί τώρα είπαν ότι έχουμε στη διάθεσή μα περιορισμένου περιορισμένους πόρους. μπορεί τα τρένα υψηλή ταχύτητα να είναι ενδιαφέροντα σε 20-30 χρόνια και γι' αυτό θέλουμε 60 τα 100 για τους σιδηροδρόμους και 20% για τους ε, δρόμους. Ε, βρίσκω ότι είναι πολύ τολμηρό από τους ε, Πολωνούς να λένε αυτό. Δεν θέλω λοιπόν περισσότερα χρήματα για τα μεγάλα έργα. Έχουμε και τα τούνελ, αποφάσεις που έχουν ληφθεί πριν πολύ καιρό και ακόμα δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Θα πρέπει να κλείσουμε το δίκτυο, να συμπληρώσουμε το, να ολοκληρώσουμε το, δίκτυο και εδώ λείπουν πολλά θέματα και γι' αυτό η ερώτησή μου είναι ε, εσείς τι πιστεύετε όταν μιλάμε για ε, διασυνοριακά ε, σημεία που έχουν καταστραφεί και αν τα... Εάν εδώ επενδύσουμε όχι το 20% αλλά το 60-70% τότε θα είναι ενδιαφέρον για τα κράτη-μέλη να πάρουν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Υπάρχουν ε, γερμανικά έργα, το Stuttgart 21, Stuttgart Ulm η διασύνδεση, ε, δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη, αλλά ε, λαμβάνει επιδότηση ένα δισεκατομμύριο από την Ευρώπη. Αλλά τα διασυνοριακά θέματα, Βερολίνο, Μπρέσλαο, εκεί δεν γίνεται τίποτα. Έχω δανό υπουργό μπροστά μου, θα μπορούσαμε πολύ γρήγορα ε, από τη Νότια Γερμανία να έχουμε ε, σύνδεση προς την Κοπενχάγη. Θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε και το ferry boat ανάμεσα στη Γερμανία και την ε, Δανία. Αυτό σε 20 χρόνια το νωρίτερο θα πραγματοποιηθεί, αλλά ξέρετε ότι στη Γερμανία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σχέδιο. Γιατί δεν προωθούνται λοιπόν τέτοια θέματα, γιατί για, για τα μικρά έργα χρειάζεται πάντα τόσο καιρό. Πάντα ε, αυτό ε, ε, ε, ε μου δημιουργεί απορίες στο Συμβούλιο. Δεν πρέπει να ε, προωθούμε το, τη μαφία των, υπο, των οικοδομών, ζητώ συγγνώμη, το, λόμπι των οικοδομών. Θα πρέπει να ε, εξετάσουμε την αποτελεσματικότητα των μεταφορών και θα πρέπει να ε, προωθήσουμε την απασχόληση. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, είναι πολύ μεγάλη η ανεργία και ιδιαίτερα των νέων. Το θέμα λοιπόν είναι πού μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Δεύτερο θέμα, η αναδιατύπωση. Βρήκαμε ένα συμβιβασμό Θέλατε παρέκκληση για ε, τα κράτη της Βαλτικής και για μια συγκεκριμένη πολωνική γραμμή. Ε, σήμερα το πρωί ελήφθη η απόφαση. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, είναι πράγματι η αλήθεια ότι η Πολωνία είπε ότι ούτως ή άλλως θα καταψηφίσουμε την αναδιατύπωση ακόμα και με την παρέκκληση αυτή και ε, έχει αναλάβει σήμερα η Πολωνία πρωτοβουλία να βρει ε, συμβιβασμό για τη γραμμή αυτή. Ε, έγινε κάτι, δεν θα το ξέρετε επειδή ήσασταν εδώ, τέλος πάντων. Όσον αφορά τους ταχυγράφους Ήδη υπόθηκαν αρκετά θέματα εδώ. Θέλουμε να μειώσουμε την γραφειοκρατία. Θα... Δεν βρίσκω πολύ καλό το ότι υπάρχουν πολλές ε, διαφορετικές ε, κατευθύνσεις όσον αφορά τα πολύ μεγάλα φορτηγά, τα monster trucks. Ε, είναι σημαντική η οδική ασφάλεια, αλλά το θέμα ότι το κόστος τελικά θα ε, το αναλάβουν τα κράτη-μέλη ε, είναι ένα θέμα και ε, δεν πριν ένα χρόνο είχε διατυπωθεί διαφορετική θέση από σήμερα και μπορεί, και η Κομισιόν πιστεύει ότι μπορεί με μια επιστολή να αλλάξει τους νόμους. Ε, η Κομισιόν αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, δεν είναι όμω ο τελικός νομοθέτης. Ε, φανταστείτε ο Μάρτιν Σούλς να γράψει μια επιστολή που να λέει ότι ε, τα πολύ μεγάλα φορτηγά δεν επιτρέπεται πια να κυκλοφορούν. Να στείλει τέτοια επιστολή προ τα, προς τα Φανταστείτε τι αντιδράσει θα υπήρχαν. Γι' αυτό πιστεύω ότι σημαντικό ως πρόεδρο του ε, Συμβουλίου να πρέπει να υπερασπιστείτε τους ε, νόμους. Συμφωνούμε ότι υπάρχει μια ε, κανονική νομοθετική διαδικασία. Ήσασταν και εσείς βουλευτής. Τι θα λέγατε εσείς αν η κυβέρνηση έλεγε ότι με ενδιαφέρει τι λέει το κοινοβούλιο, εμείς θα, το, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ε, διαδικασίας. Δεν ε, μπορούμε να ε, δεχτούμε κάτι τέτοιο, διότι θα αποτελέσει και προηγούμενο για άλλες αποφάσεις. Θα είμαι τώρα πάλι θετικός. Ήταν πολύ θετική η πρωτοβουλία σας και το, η, η, η διάσκεψη που, οργανώσανε, οργανώσατε για το EFTMS. Ε, με το πρόγραμμα αυτό το 20 25% της ε, κατανάλωσης ενέργειας ε, μπορεί να εξοικονομηθεί με τα ηλεκτρονικά φρένα. Αυτό είναι θετικό. Με τα ηλεκτρονικά φρένα θα έχουμε και μείωση του θορύβου κατά 10 δεσιμπέλ. Μόνο με δύο θέματα δηλαδή ε, που έχουν να κάνουν με τους ε, σιδηροδρόμους, ε, δηλαδή και με την εξοικονόμηση της ενέργειας και μείωση των δεσιμπέλ, έχουμε λόγους να εφαρμόσουμε το μέτρο αυτό. Όσον, αφορά το πακέτο των ε, αεροδρομίων, αναφερθήκατε σε αυτό, δεν έχουμε προχωρήσει πολύ στο θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ κακό ότι η Κομισιόν λέει ότι θέλουμε να αποφασίσουμε ε, εάν ε, είναι λογική η μείωση της λειτουργίας. Πολύ σωστά δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό και το Συμβούλιο το είπε αυτό. Για, για, φανταστείτε να λέει ότι θα σταματήσουν οι νυχτερινές πτήσεις ε, στη Φραγκφούρτη. Ε, δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πιο αντιευρωπαϊκή ρύθμιση. Ε, δεν αναφερθήκατε όμως στο σύστημα εμπορίες εκπομπών στις αερομεταφορές. Ακούσαμε τις αντιρρήσεις Ηνωμένων Πολιτειών ε, και Κίνας ε, και μάλιστα οι αντιρρήσει ε, που ακούστηκαν ήταν ότι φοβήθηκαν ότι το μέτρο αυτό θα εφαρμοστεί και στις ναυτιλιακές εργασίες. Και επίσης, από ό,τι άκουσα ο Γερμανό ομολογός σας, είπε ότι οι Κινέζοι ακύρωσαν τις παραγγελίες Airbus. Αυτό ήταν μια απειλή, διότι Ξένα ε, έκαναν την παραγγελία αυτή. Τρέχει λοιπόν το θέμα αυτό, αλλά ε, η θέση του Συμβουλίου ε, ποια είναι. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτό. Άλλωστε το δικαστήριο το έχει επιβεβαιώσει. Όσον αφορά τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους. Ε, πολύ καλό αυτό και οι κοινωνικές ε, συνθήκες παίζουν ρόλο. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό. Σας ευχαριστώ για την ε, συνεργασία. Ελπίζω ότι ακόμα και όταν δεν θα είστε πια προεδρεύον του Συμβουλίου θα συνεχιστεί η συνεργασία μας. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Έχετε 30 λεπτά ξεχαστικά. Δεν χρειάζομαι καν 30 δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. Στην αποστολή της Τραν Ε, ήσασταν ε, παρόν και ε, πήρατε θέση και πιστεύω ότι αυτό ήταν πολύ θετικό από πλευρά σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Τσίλε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τη Δανική Προεδρία και τον κύριο Υπουργό για τα όσα επιτυχάτε κατά την Προεδρία σας στον τομέα των μεταφορών. Πρώτα απ' όλα σημειώστε τεράστια πρόοδο για το, στο μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη και στις κατευθυντήριες γραμμές ε, του ΤΕΝΤΗ. Συγχαρητήριο. Λοιπόν, γι' αυτό η πρόταση της Κομισιόν παρέχει ένα νέο νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των ε, δικτύων μεταφορών ε, σε διάστημα 7 ετών. Καλό είναι να έχουμε λοιπόν το κατάλληλο χρηματοδοτικό μέσο για το Connecting Europe. Χρειάζεστε αυτό το χρηματοοικονομικό μέσο, διότι το εύρος της ε, χρηματοδότησης έχει μειωθεί στο απαραίτητο ελάχιστο. Χρειαζόμαστε να είναι αυτό το μέσο αποτελεσματικό. Είναι αυτό δυνατό, ορισμένα κρατημένοι. Απλά δεν έχουν κονδύλια να διαθέσουν σε υποδομές μεταφορών. Σκέφτομαι τώρα και τα ζητήματα συνοχής 10 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Συνοχής θα πάνε στο μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη, στο Connecting Europe. έχετε όμω 30% συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τους διαδρόμους. Αυτό δεν θα αρκέσει ώστε αυτά τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να επιλύσουμε. Επίσης, οι χώρες οι οποίες πιέζουν για μείωση του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορισμένες φορές ε, μιλούν για μεγαλύτερη δημοσιονομική ενοποίηση. Αυτό φαίνεται να είναι δύο αντικρουόμενα πράγματα. Εφόσον έχουμε πολιτική ένωση στην Ευρώπη, χρειαζόμαστε σίγουρα μεγαλύτερο προπολογισμό ώστε να βοηθήσει να αναπτυχθούν οι περιφερειακές ε, χώρες που βρίσκονται σε ε, λιγότερο καλή θέση όσον αφορά τις υποδομές των μεταφορών. Όσον αφορά τώρα τις θαλάσσιες μεταφορές, στο ζήτημα της ε, σαφήνειας. Η ομάδα μας το έχει μελετήσει πολύ. Ευχαριστούμε για τα επιτεύγματά σας σε αυτήν την τομέα. Όσον αφορά την εκπαίδευση των ναυτικών, επίσης, το τρίτο σημείο για την αναδιατύπωση της δέσμης μέτρων για τους ιδεοδρόμους πρόκειται για κάτι δύσκολο και έχετε επιτύχει κάποια πράγματα εκεί. Αυτή η επιστολή όμως ε, που εστάλει από την Προεδρία θα έλεγα ότι εάν θεωρούμε ότι η νομοθεσία προωθεί την ανταγωνισμό μεταξύ των εταιριών στην Ευρώπη, τότε βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Εάν όμως ε, εμπλακούν και τρίτες χώρες στο δικτύο μας, τότε μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Είτε μιλάμε για μια πολωνική γραμμή, ένα πολωνικό δρομολόγιο, είτε για γραμμές ε, στις χώρες της Βαλτικής. Ε, υπάρχει, υπάρχει ξέρετε ένα σύστημα μέσω της ε, ε, Ρωσίας μέχρι τη Βόρεια Κορέα. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε για αυτή την εξαίρεση. Οι συμβασμοί χρειάστηκαν πολύ καιρό στο Κοινοβούλιο. διότι οι ρυθμιστικές αρχές για τη Βαλτική χρειάζονταν την δυνατότητα να αναλάβουν δράση σε σχέση με φορείς ε, τρίτων χωρών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις χώρες μας, τόσο πολύ που δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς αυτό στην νομοθεσία. Αυτό που ακούσαμε μόλις να λέει η κυρία Μάισνερ σημαίνει ότι δεν θα μπορέσετε να αποφασίσετε μόνοι σας για το ενίο ευρωπαϊκό ουρανό, ούτε εμείς μπορούμε. Ποιος θα το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ η κυρία Φώστερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Προεδρία. Ε, θέλω να προσθέσω ορισμένα στοιχεία που αφορούν την άποψη της μας ομάδας. Όταν είπατε ότι ο υπουργό δεν μπόρεσε να έρθει, ο αρμόδιος για, το, για τον ε, τομέα αυτό, όλοι μαζί προσπαθούμε να προβληματιστούμε κάπως καλύτερα από τα όσα είπε για την αεροπλοή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να τα πάμε κάπως καλύτερα και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι οι τρίτες χώρες θα συμφωνήσουν και όλοι λοιπόν γύρω από ένα τραπέζι θα αποφασίσουν το καλύτερο για το μέλλον. Να μην επισέλθω όσα έδειξε ο συνάδελφος για το ETS, ο συνάδελφος των Πρασίνων. Ξέρουμε ότι η κατάσταση εκεί είναι τραγική και τα πράγματα δεν προχωρούν πολύ καλά, όμως ε, συμφωνώ ε, για όσο για την πειρατεία, πολύ σημαντικό το ότι αντιμετωπίζονται τα προβλήματα εκεί. Τώρα κάτι άλλο, όσον αφορά τους ταχογράφους. Είναι πολύ σημαντικό, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών και βέβαια ε, αυτό που θέλουμε όλοι είναι να λειτουργεί ευρυθμό το σύστημα και όλοι συμφωνούν με το σκοπό αυτό. Όμως έχουμε διαφορετικές ε, λεπτομέρειες που ανακυβλούν σε σχέση με τον τρόπο που θα φτάσουμε στον κοινό σκοπό. Και να δούμε το ότι ορισμένα κρατημέλη έχουν τις κατάλληλες υποδομές και δεν χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Οπότε δεν χρειάζεται να τα εναρμονίσετε όλα. Απλώς να εξασφαλίσετε ότι τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για το ότι κάνουν. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Γαλιλαίου και της υποδομής, μεγάλη μας χαρά είδαμε ότι το θίξατε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτού του είδους οι υποδομές να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Είναι σημαντικό αυτό ε, να ε, τηρούνται τα, τα επισχήματα κράτη-μέλη και να δούμε κατά πόσον μπορούμε να, να καταφέρουμε να μην χάσουν το τρένο της τεχνολογίας. και για κάποια στιγμή πλοήγησης παγκόσμια με δορυφόρο. Είμαι η συγγήτρια και επίσης όσον αφορά τον ενίο ουρανό και το ΦΑΠΣ επίσης, ε, Ιρλανδία και Δανία έχουν κάνει πρόοδους, αλλά μάλλον ψωδρόμηση έχουμε στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά θα πρέπει κάτι να κάνουμε όσον αφορά την, την υπερβολική κυκλοφορία, να έχουμε καλύτερη διαχείριση στην αεροπλοεία και το θέμα είναι το πώς δεν θα μετακυλείται το κόστος ή τέλος πάντων οι περικοπές στον καταναλωτή και άρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να σημαίνεται πρόοδος. Ένα από τα θετικότερα είναι ότι προσπαθήσαμε να... Η Δανέζικη Προεδρία όντως βρήκε τη συνένεση για το PNR Μα πήρε μια δεκαετία, αλλά τελικά καλά τα πήγατε, τα βρήκαμε. Τρώσαν φρέτα σφαγιαλέ στα αεροδρόμια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα στο Κοινοβούλιο και όχι, δεν είναι ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει χαλαρότητα. Στο αντίθετο, με τίποτα θέλουμε χαλαρότητα. Όμως το θέμα είναι τι είδου μηχανήματα θα υπάρχουν, ε, αν θα υπάρχει ε, κάποιο ακτινοβολία, ε, υπάρχουν κάποια συστήματα με ήχους, υπερήχους που είναι αλλακτική λύση. και δεν μπορείτε να, να επιβάλλετε στα μελη το τι θα χρησιμοποιήσουν γιατί πολλές φορές η επιστημονική τεκμηρίωση λέει τα εντελώ αντίθετα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα επομένω τέλο πάντων. Εν κατακλείδιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Δανεισική Προεδρία. Ξέρουμε ότι επίσης και η Κυπριακή Προεδρία παρακολουθεί τα θέματα της αεροπλοείας, έρχονται πάντα εδώ στις συνεδριάσεις πάμε καλά, κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν πιο διάφανα, δεν χρειάζονται τίποτα ανατρεπτικές μεγάλες αλλαγές. Η Δανία, η πήγε με την Προεδρία πάντως πάρα πάρα πολύ καλά. Κύριε Φώστερ, ευχαριστούμε. Κύριε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Δανέζικη Προεδρία πιο δύσκολο έργο ήταν η προώθηση της αναδιατύπωσης, αλλά ήδη ακούστηκαν αρκετές παρατηρήσεις γι' αυτό. Η Δανία δεν είναι μεγάλο κράτος σε σιδηροδρόμων, είναι όμως σημαντικό ναυτιλιακό κράτος. Ε, εμένα είπα, ε, εγώ προέρχομαι από πολύ κοντά από τη Βαλτική και Ε, είχαμε εξελίξεις που δείχνουν πόσο σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των ναυτικών, ε, να βελτιώσουμε την ασφάλεια στα πλοία. Να χρησιμοποιούμε το καλλιλέο στο μέλλον ε, για την πλοήγηση των πλοίων. Η Βαλτική είναι κλειστή θάλασσα και έχει την μεγαλύτερη ε, κυκλοφορία πλοίων στον κόσμο. Ο Ντομινίκ Ρικέ είναι εισηγητής για τα δεξαμενόπλια διπλού κήτους. Εάν κοιτάξουμε πόσο πετρέλαιο μεταφέρεται ε, στη θάλασσα και ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τις μεταφορές αυτές, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σύντομα με το θέμα των δεξαμενόπλειων ε, διπλού Εκατομμύρια τόνους ε, πετρελαίου μεταφέρει ε, η Ρωσική Ομοσπονδία σε όλο τον κόσμο. Σας καλώ λοιπόν και μετά την Προεδρία σας να φροντίσετε να εφαρμοστούν αυτές οι κοινέ πρωτοβουλίες. Όσον αφορά τις περιοχές ελέγχου το 2015 θα ε, τεθούν σε ισχύ οι κανόνες ε, σχετικά με τα όρια του θείου Ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες χωρίς να στρεβλωθεί ο ανταγωνισμός. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, συζητήσαμε ε, και εδώ και ξέρω επίσης ότι το συζήτησε η Προεδρία σας. σα ευχαριστώ πάντως για τις επιτυχίες σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ δεν ζήτησε κάποιος άλλος τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, ακούσατε τις απόψεις των μελών αυτής της Επιτροπής Μεταφορών που εκφράζουν ε, ανησυχίες ε, ε, παρόμοιες για τα διάφορα συστήματα. Επίσης εξέφρασαν μια έντονη αναγνώριση της δράσης σας ε, δράση που αφορούσε ορισμένε φορέ ευαίσθητα θέματα, όχι μόνο για τις μεταφορές αλλά και σε άλλα επίπεδα. Ε, σίγουρα χρησιμεύσατε ως σημείο καμπής ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όλοι οι βουλευτέ εξέφρασαν ανησυχίε όσον αφορά τα δίκτυα και το μηχανισμό συνδέοντα την Ευρώπη, που συνεχίζει να αποτελεί ένα ζήτημα που θα απασχολεί στο μέλλον. Αναγνωρίστηκε επίσης η συμβολή σα στην αναδιατύπωση ε, του κειμένου για του σιδηροδρόμου καθώς και για το ζήτημα που αφορά τα μεγάλα φορτηγά. Σα δίνω λοιπόν τον λόγο κύριε Υπουργέ ώστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακούστηκαν και να μας πείτε τα συμπεράσματά Σα Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ε, και προς τον ε, συνάδελφο Σόν ε, που θα του τα μεταφέρω. Υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά θα ήταν πολύ δύσκολο και δεν έχω και τον χρόνο να απαντήσω σε πολλά από αυτά που είπατε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να αναφερθώ σε κάποιες από τις γενικές παρατηρήσεις που έγιναν. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας όσον αφορά ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το CEF. Δεν έχουμε ολοκληρώσει το θέμα αυτό ακόμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ε, Τραν θα ε, συμμετάσχουν πολύ. Αλλά είχαμε μια γενική προσέγγιση από τους ε, υπουργού μεταφορών της Ευρώπης. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό οι υπουργοί μεταφορών να υποδείξουν πού θα πρέπει να υπάρχουν οι βασικοί διάδρομοι για τη μεταφορά επιβατών και ε, αγαθών στην Ευρώπη στο μέλλον. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τη δική μας δουλειά, δηλαδή να δούμε πού θα έχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία με, τις, ε, με την ε, διασφάλιση καλών μεταφορών, τότε δεν μπορούμε και εμείς να πάμε στους υπουργούς οικονομικών και να πούμε ότι θέλουμε χρήματα. Αν θέλουμε χρήματα θα πρέπει να μπορούμε να απαντήσουμε τι τα θέλουμε. Και γι' αυτό Πιστεύω ότι με τη γενική προσέγγιση όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα και το CEF ε, έχουν κάνει ε, τα δικά τους μαθήματα και μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια της συζήτησης και να δούμε πού θα καταλήξουμε όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το διάστημα 2014 με 2020. Πάντως εγώ χαίρομαι που νιώθω ότι οι Υπουργοί Μεταφορών έκαναν τη δική τους δουλειά όσον αφορά το πακέτο αεροδρομίων. Αυτό που μας απασχόλησε πολύ ήταν να δώσουμε συνέχεια ε, στις, ε, στις εργασίες. Ε, ιδιαίτερα μας ενδιέφεραν οι υπηρεσίες εδάφους και ο θόρυβος. Δεν έχουμε συζητήσει τα σλότ ε, κατά τη διάρκεια της θέση ε, προ δηλαδή κατά τη διάρκεια της δικής μας της Προεδρίας. Ε, χαίρομαι όμως που καλύψαμε δύο από τα τρία αυτά θέματα. Τώρα παραδίδουμε την σκητάλη και στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι λοιπόν που τα καταφέραμε. Όσον αφορά τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, θυμάμαι ότι όταν σας παρουσίασα τη Δανέζικη Προεδρία, Πολλοί από τους βουλευτές της Επιτροπής ΕΤΡΑΝ ε, με ρώτησαν για το θέμα αυτό. Δεν έχουν γίνει πολλά στο θέμα αυτό δεν, ε, να πω στην κυρία Μάισνερ ότι δεν λάβαμε σχετικές προτάσεις, αλλά συμφωνώ ότι θα πρέπει να πάρουμε στο σοβαρά το θέμα αυτό και ε, θα ε, βοηθήσουμε στην επεξεργασία του θέματος αυτού, αν έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε αυτό, κατά διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Δεν θέλω να ανακατευτώ στην συζήτηση ανάμεσα στην Επιτροπή σας και την Κομισιόν όσον αφορά την νομοθεσία. Αλλά μπορώ να σας ε, μιλήσω για τις δανέζικες εμπειρίες, διότι τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουμε ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό. Εμένα με απασχόλησε το θέμα, επειδή βλέπω ότι μπορούμε να κερδίσουμε και από οικονομικής πλευράς και από οικολογικής πλευράς. Δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα πότε θα πρέπει να ε, έχουμε νομοθεσία και πότε όχι, απλά έχω την ε, γενική μου αυτή θέση που έχει να κάνει με την οικονομία και την οικολογία. Στον κύριο Γκρός να πω ότι όσον αφορά το κοινωνικό dumping στις μεταφορές, αυτή είναι μια συζήτηση ε, η οποία βλέπω να γίνεται όλο και πιο ανησυχητική και να ε, εστιάζεται και περισσότερο. Και στη Δανία γίνεται η συζήτηση αυτή και εμείς οι αρμόδιοι υπουργοί, οι αρμόδιοι πολιτικοί θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο θέμα αυτό τα επόμενα χρόνια στην κυρία Μάισνερ να πω ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική είναι ένα θέμα για το οποίο δεν γνωρίζω τίποτα. Νομίζω μάλιστα ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος. Δυστυχώς δεν μπορώ να ε, σας απαντήσω στο θέμα αυτό. Ε, πάντως ε, εγώ χάρηκα που ε, συνάντησα την ε, Επιτροπή Τραν ε, κατά τη διάρκεια της αποστολής της. Ήταν πολύ καλή η επίσκεψη αυτή στον κύριο Κράμερ ε, να πω ότι ζητάτε αναλύσεις. Θα πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό, διότι συχνά βλέπω στο τέλος των ε, διασυνοριακών έργων ε, και των μικρών έργων να μην ε, να μην ε, έχουν την προσοχή του κόσμου, ε, ενώ θα μπορούσαν να δώσουν ευρωπαϊκή προστιθεμένη αξία. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε. Και νομίζω ότι αρκετοί είπαν, νομίζω ότι και η κυρία Φώστερα αναφέρθηκε στο θέμα των περιβαλλοντικών τελών και την συζήτηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Ε, ε, σύντομα ενημερώθηκαν οι Υπουργοί ε, Μεταφορών, αλλά νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι αρμοδιότητα των Υπουργών που είναι υπεύθυνοι για την αλλαγή του κλίματος. Δανέζα Υπουργό εκεί είναι η κυρία Χέντεκορτ. Είναι λοιπόν κάτι που δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ στον κύκλο των Υπουργών Μεταφορών. Η κυρία Φώστερ αναφέρθηκε και στον Καλλιλέο. Συμφωνώ με τις ερωτήσεις της. καθώς και με το ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά στον τομέα αυτών. Να πω στην κυρία Φώστερ ότι η δανοσουηδική ε, συνεργασία λειτουργεί πολύ καλά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο με τις άλλες ε, χώρες ε, της Βορείου Ευρώπης για να έχουμε, περισσότερο, να έχουμε καλύτερο έλεγχο στον ουρανό της Βορείου Ευρώπης. Και Κύριε Πρόεδρε, δεν ε, μπόρεσα να απαντήσω πολύ αναλυτικά στις ε, πολλές ερωτήσεις που τέθηκαν. Προσπάθησα όμως να σας δώσω κάποιες γενικές απαντήσεις. Σας ευχαριστώ και πάλι για τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας, για το έργο σας και για την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις που δώσετε στις ερωτήσεις μας σήμερα. Εδώ διακόπτεται η συνεδρίμαση μας. Θα συνεχίσουμε στις 3 η ώρα για τα υπόλοιπα θέματα. thank you for coming and taking more time than expected. It's okay. We were running late with the rollers. yeah. this can happen in Parliament. Yeah, Yeah, yeah.